Eh, λοιπόν, συνάδελφοι, ε, ας αρχίσουμε σιγά σιγά. Έχουμε μερικές ε, χιλιάδες τροπολογίες να ψηφίσουμε. Καταρχάς να δούμε τη μέση διάταξη. Στα νέα της Επιτροπής μας μπορείτε να διαβάσετε ότι πρέπει να αλλάξουμε τη μέση διάταξη. εμείς ως Κοινοβούλιο λάβαμε το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης του Συμβουλίου για την αναθεώρηση του κανονισμού της Όλαφ. Θα πάει και στην Ολομέλεια και βάσει του κανονισμού μας θα πρέπει να το εγγράψουμε ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας αλλά επειδή έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες προτείνουμε αυτό το θέμα να το συζητήσουμε αύριο το απόγευμα στο σημείο 58 παρακαλώ της ημερήσιας διάταξης και υπολογίζουμε να γίνει αυτό γύρω στις 5 το απόγευμα. Κάτι άλλο που συνδέεται λίγο με αυτό, στο μεταξύ λάβαμε και επιστολή Ε, του Προέδρου της ε, Εποπτικής ε, Επιτροπής που δηλώνει, επιβεβαιώνει μάλλον την παρέτηση της Ρίτα Σέμπρη που παρετήθηκε από την Λόγο Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι μετά την υπόθεση Ντάλι, το σκάνδαλο, έγινε μια έκθεση της Επιτροπής αυτής ε, για την έρευνα που έκανε η Όλαφ και μετά από πίεση και της δικής μας Επιτροπής. Στο μεταξύ έχουμε την έκθεση αυτή, την έχουν στείλει στο Κοινοβούλιο. Ακόμα μπορούν να τη δουν ε, ορισμένοι, είναι σε κλειστό κύκλο, με μονομένοι βουλευτές. Και ζήτησε ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής της Εποπτικής επειδή έχει δημιουργηθεί σάλος, ε, να έρθει αύριο στην Επιτροπή μας για μια γενική ενημέρωση για όλες τις έρευνες που διεξάγει η Επιτροπή ε, σε σχέση με τις έρευνες που κάνει και η Όλαφ, η Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης. Να καλέσουμε τον κύριο Τενχόφ δηλαδή, ε, πριν το σημείο της Όλαφ, ε, πριν το 58, πάλι αύριο το απόγευμα κατά τις 5. Συμφωνείτε λοιπόν με αυτή την αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω παρά συμφωνία λοιπόν. Εγκρίνεται με τις αλλαγές αυτές η ημερήσια διάταξη. Έχω μερικές μόνο ανακοινώσεις περιορισμένες, τις οποίες θα βρείτε όλες συνοπτικά ε, στο Cont News, ε, συνεδρίαση της άλλης εβδομάδας της Δευτέρας ακυρώνεται. Ε, ήταν εφεδρική, την είχαμε βάλει έτσι μήπως χρειαστεί. Ε, οπότε μπορούμε να έχουμε ελεύθερο αυτό το απόγευμα. Και κάποια θέματα επίσημα. Καλωσορίζουμε τη Φάνη Προύξ. Ε, καινούργια στη γραμματεία έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Δεν τη βλέπω, δεν τη γνωρίζω κιόλας για να τη δω. Καλωσορίσατε κυρία Μπρούξ και ελπίζουμε ε, σε μια πρόσκοπτη και καλή συνεργασία. Ο κύριος Πιότρ Μπαρτοσίβιτς Μαλίκη, πώς το προφέρουν αυτό, ε, έχει εργαστεί ε, για λίγο διάστημα στην Επιτροπή μας και τώρα μετατέθηκε στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Καλή σταδιοδρομία λοιπόν και καλή τύχη στα καθήκοντά του. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μου. Και τώρα μου λέγει η Κάρμεν ότι δεν θα έρθει ο ίδιος ο κύριος Στενχόφ αύριο, αλλά ο πρώην συνάδελφός μας, ο κύριος Μπέος, για να μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Τίποτα άλλες παρατηρήσεις έχουμε, ο Γιάννης Γκάιερ. Μια ερώτηση μόνο. Μπάρτ, ε, πόσο χρόνο θα πάρει δηλαδή αυτό το σημείο της ημέρησιας διάταξης με τον συνάδελφο Μπέος. Είναι πάρα πολύ φορτωμένη η ημερήσια διάταξη. Ε, πρώτη φορά έχουμε τόσο βαριά ημερήσια διάταξη. Και ε, έχουμε να συζητήσουμε και τα θέματα της εποπτικής αρχής της Όλαφ και σύμφωνα με την εμπειρία μας αυτά δεν διεκπαιρεώνται μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας. Έχω μεγάλη ανησυχία μην υπονομεύσουμε την ίδια μας ημερήσια διάταξη για μια τέτοια συζήτηση με την Επιτροπή Εποπτείας Όλαφ. Τον ξέρω πολύ καλά το Herbert και χαίρεται να τα λέει και πάρα πολύ αναλυτικά. Και θα μας πάρει μια ώρα η συζήτηση μαζί του. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει στην παρούσα ε, συνεδρίαση αυτή η συνάντηση. Γένς, ε, όπως και να έχουν τα πράγματα, θα έχουν τελειώσει όλες οι ψηφοφορίες, ελπίζω θα ψηφίζουμε ε, συνεχώς μέχρι να τελειώσουν όλες οι ψηφοφορίες για τις απαλλαγές. Αυτές θα πρέπει να έχουν λήξει. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν όλων των ψηφοφοριών, τι έγινε, δεν υπάρχει διερμηνία από τα Ολλανδικά και βέβαια υπάρχει. Λοιπόν, εμ, Ελπίζω λέγω να έχουν τελειώσει όλες οι ψηφοφορίες και κανονικά είμαστε εντάξει για τις απαλλαγές. Μετά θα συνεδριάσουν 4 με 5 οι συντονιστές. Είχαμε προγραμματισμένη συνεδρίαση των συντονιστών η οποία καταργείται. Έχουμε λοιπόν ένα χρονικό περιθώριο. Και ακούω τη συζήτηση, μου λέγει η γραμματεία, με τον κύριο Μπέος. Θα διαρκέσει 30 με 45 λεπτά. Δηλαδή κανονικά προλαβαίνουμε γιατί ε, είπαμε ματαιώθηκε η συνάντηση, η συνεδρίαση των συντονιστών. Εντάξει, διασκεδάστηκαν οι φόβοι σας. Η κυρία Γκρέσλε, ως εισηγήτρια σας υπόσχομαι να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Δεν το κατάλαβα αυτό, λέει ε, ο κύριος Στάς. Μα εγώ είμαι εισηγήτρια, λέγω, για το σημείο 58 και σας υπόσχομαι να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Μάλιστα, το σημειώνουμε και αυτό. Ποιος συνάδελφος θέλει το λόγο. Ο κύριος Μπράντμπορν. Έχω ένα διαδικαστικό, δεν ξέρω θα πρέπει να το πω τώρα, πριν αρχίσουμε τις ψηφοφορίες για όλες αυτές τις διαδικασίες συναλλαγής, ε, ε απαλλαγής. Ε, πότε να το πω αυτό το διαδικαστικό μου. Μια στιγμή να σας πω, λέει ο Πρόεδρος. Κανονικά θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα όλες τις εκθέσεις για την απαλλαγή. Εάν έχετε διαδικαστικό, να το πείτε τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, την περασμένη εβδομάδα, αφού έφυγα από το Στρασβούργο, δέχτηκε εδώ το γραφείο μου στις Βρυξέλλες ένα τηλεφώνημα από διευθυντή ενός οργανισμού για τον οποίο ψηφίζουμε σήμερα την απαλλαγή. Τι έλεγε λοιπόν αυτό το τηλεφώνημα του διευθυντού. Δεν θα σας πω τον οργανισμό γιατί είναι θέμα αρχής. Ήταν να αμφισβητήσει και να ρωτήσει γιατί έχω βάλει εγώ τροπολογίε σε αυτή την έκθεση για την απαλλαγή του οργανισμού. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι είναι σωστό τρόπο συμπεριφορά αυτό ε, για ένα ανώτατο υπάλληλο ε, σε ένα οργανισμό. Ε, δεν είναι αρμόζουσα αυτή η συμπεριφορά και επίσης δεν δέχομαι ως βουλευτής να με ρωτάει ένας υπάλληλο γιατί κάνω τροπολογίες για εκθέσεις ή έγγραφα της Επιτροπής. Διαμαρτύρομαι εντόνως. Δεν είναι σωστή η συμπεριφορά ούτε διαδικασία όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον ε, για να λειτουργούμε ε, σωστά στα θεσμικά όργανα και ελπίζω να συμφωνήσει και η Επιτροπή μας ότι είναι τελείως ανάρμοστο ε, να ρωτάνε ένα βουλευτή ε, γιατί έκανε τροπολογίες. Μα αυτή είναι η ουσία της δουλειά μας. Eh, er Ευχαριστώ. Ε, θέλει κανείς άλλο το λόγο? Ο κύριος ε, Ρούμπιχ, όχι ο κύριος Ρούμπιχ, λάθος. Είδα να συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι την ώρα που μιλούσατε. Ε, το σημειώνουμε. Σας προσέγγισαν όχι μόνο σας και κάποιους άλλους και εγώ προσωπικά έχω αυτή την εμπειρία δεχτήκαμε κρούσεις και θα πρέπει πραγματικά να, να το αντιμετωπίσουμε με το σωστό τρόπο. Έχετε απολύτως δίκιο. Πριν αρχίσουμε τις προφορίες, έχουμε άλλες παρατηρήσεις. Όχι. Ωραία. Σημείο 3. Απαλλαγή για την Επιτροπή. Η είναι ο κύριος Γιάνς Γκάιερ. Θες να πεις τίποτα Γιάννη εισαγωγικά, όχι, όλα είναι ξεκάθαρα. Καλώ ας ψηφίσουμε λοιπόν. Να ετοιμάσουμε τα χαρτιά μας. Εγώ πρέπει να προσέχω ταυτόχρονα δύο έγγραφα. Κυρία Χέρτσοκ, έρχεται η κάρτα μου. Παρακαλώ για λίγα λεπτά δεχτείτε να ψηφίζω διανατάσεις στους χειρός. Μάλιστα. Ωραία, θα σας παρακολουθούμε πώς θα ψηφίζετε και θα μετράμε αντίστοιχα την ψήφο σας. Είστε όλοι έτοιμοι. Πάμε, είναι μεγάλη ψηφοφορία. Παράγραφος 1, η τροπολογία 1 του κυρίου Μπράτμπον. Υπέρ. Κατά, αποχές. Απορρίφτεται. Η τροπολογία 2 του κυρίου Οντί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τότε θα ψηφίσουμε την πρόταση απόφαση όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία τώρα ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Να προσθέσουμε στους 21 υπέρ και μία ψήφο. 22-4 συγκρίνεται. Και προχωρούμε. Παράγραφος πρώτη τροπολογία 3 του κυρίου μπραντμον και Τσαρνέσκι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απόρριψες. Μια προφορική τροπολογία του Γέντς ε, γαιερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το σύνολο. 21 υπέρ 5 κατά. Κυρία Χέρτσοκ, να μας πείτε όταν φτάσει η κάρτα σας. Ε, μη σας μετράμε. Ε, και προχωρούμε. Παράγραφος πρώτη, τροπολογία 4 των ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και πάλι προφορική του κυρίου Γκάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά το σύνολο λοιπόν της πρότασης. Άρχιτε ψηφοφορία, πέρας. Άνοιξε ψηφοφορία, ναι. Έκλεισε κιόλας. 21-5 εγκρίνεται. τροπολογία 5 στην παράγραφο 1 και πάλι η Bradburn και Τσαρνέκη είπε κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική του Γκάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο. Πέρασα. Αποτέλεσμα 22 υπέρ, 4 κατά εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία. Η παράγραφος 1 πάντα, 6, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία του κυρίου Γκάιερ υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πέμπτη ψηφοφορία. Πέρας. Είκοσι ένα υπέρ. Πέντε κατά εγκρίνεται. Η επόμενη ψηφοφορία έκτη. Στην πρώτη παράγραφο τροπολογία 7. Μπραντ Τσανέκη υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία Γκάιρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο πέρας 22 υπέρ 5 κατά εφταση έφτασε η κάρτα. Ωραία, 21, 5. Το 7 για τον εκτελεστικό οργανισμό για τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα, παράγραφος 1, τροπολογία 8, με τους ίδιους συντάκτες, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, ε, προφορική γκάιερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ε, ηλεκτρονικά τώρα την ε, πρόταση που βρίσκεται στη σελίδα 8. Πέρασε. Εγκρίνεται 22-4. Πάμε στην επόμενη σελίδα παριθμόν 9. Πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών. Ορίστε. Α, δεν πρέπει να το ψηφίσουμε γιατί έχουμε δώσει ήδη απαλλαγή. Οπότε ε, καταπίπτει η τροπολογία του κυρίου Μπράτπον, η ηλεκτρονική όμως όχι. Ούτε ηλεκτρονική. Ωραία, γυρίζουμε σελίδα λοιπόν. Σελίδα 10. Α, τώρα ερχόμαστε στο ψήφισμα. We close the accounts and we grant the discharge. Okay? Toch eventjes check voor de zekerheid. Λοιπόν, πάμε στο ψήφισμα. Στη σελίδα 10. Παράγραφος πρώτη, η τροπολογία 10, πίπερ, υπέρ, κατά, αποχές, θα το ελέξουμε γιατί είναι πολύ ασαφές. Πέρασε, αν ψηφίσατε όλοι. Και αποτέλεσμα εγκρίνεται 14 υπέρ 12 κατά. Παράγραφος 1, σημείο α, τροπολογία 11 του κυρίου Γκάιερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 καταπίπτει. 13, δικιά μου. Συμβατή με την 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1α νέα δική μου 14 με την προφορική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 15 του κυρίου Οντή με την προφορική τροπολογία του ΕΛΚ πάλι υπέρ. Κατά. Άποχες είναι πολύ μικρή διαφορά και χρειάζεται έλεγχο. Λοιπόν, αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Πέρας. 12 υπέρ, 14 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 16 Γκάιερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Η 17 της κυρίας Μακοβέη. Ψήφιπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, να επιστρέψουμε λίγο στην τροπολογία 15 του κυρίου Οντή. Απερίφθη η, προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Πρέπει να ψηφίσουμε όμως το αρχικό κείμενο. Άρα ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και το αρχικό κείμενο. Λοιπόν, τροπολογία 18 του κυρίου Γκάιερ. Στην παράγραφο 1 σε ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. because the compromise replaces many amendments. And Amendment 94, you can find it? Yes, that is on page... first is, Η πρόταση είναι τώρα εδώ να ψηφίσουμε πρώτα τη συμβαστική 1 διότι καλύπτει και αυτή την τροπολογία. και η, τροπολογία 94 στη σελίδα 16. Αυτό προτείνεται να ψηφίσουμε πρώτα, γιατί καλύπτονται πολλές τροπολογίες. Λοιπόν, ψηφίζουμε στην σελίδα 16 την 94 ως συμβιβαστική. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Επιστρέφουμε τώρα λοιπόν σε σελίδα 11 και είμαστε στην τροπολογία 20 της κυρίας Γκρέσλε και δική μου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 21 Γκρέσλε και Στάς υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 22 Γκρέσλε και δική μου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος πρώτη σε ένα καινούριο. Νέα, 23 του κυρίου Πίπερ, συμβιβαστική τροπολογία εδώ, υπαριθμών 2. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24, τροπολογία του κυρίου Γκάιερ υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 25. Μπράτβορν και Τσαρνέσκι. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρή διαφορά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Την τροπολογία 25 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Mm. Δεν είναι και τόσο μικρή διαφορά. 17 υπέρ, 10 κατά. Εγκρίνεται. 26 τι κάνει, κατά πίπτη. Όχι. Τι ψηφίζουμε. Είναι δική μου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 του κυρίου Γκάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 δική μου συμβατή με την 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και ερχόμαστε τώρα στη σελίδα 12, η τροπολογία 29 της κυρίας Παναγιώτοβα. Οπέ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 30 του Γκάιερ. πέ, Κατά. Εγκρίνεται. Η 31. Γιάννης Γκάιερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32. Γκάιερ υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 33. Γκάιερ υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 34. τη κυρία Πατράου Νέβης. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 35. Γκάιερ υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η 36 Γκάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ερχόμαστε στην 39 του Πίπερ με προφορική τροπολογία του ΕΛΚ υπέρ κατά Άποχες. Εγκρίνεται. 40 πι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 41 γκάιερ υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 42 γκάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 γκάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 Γκάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 δική μου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε σε 13, 47 δική μου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 48 του ΠΥΠΕΡ με την προφορική τροπολογία του ΕΛΚ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 49 δική μου με προφορική τροπολογία του ΕΛΚ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 50. Μπραντ Τσαρνέκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51. Γκάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 γκάι ριπέρ κατά αποχές έλεγχος επαλήθευση δηλαδή 52 52 52 εδώ λίγη ψηφοφορία υπέρ 8 κατά 19 απερίφθη. 53 δική μου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 πάλι δική μου συμβαστική 3 υπέρ συμβαστικής 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 δική μου πάλι με προφορική τροπολογία ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 γκάιερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 δική μου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. 58 Μπράντμπουρν Τσαρνίκη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αυτή. Θέλετε παρήθευση επαλήθευση 58. Λίγη, λίγη ψηφοφορία. Α, εγκρίνεται. Τώρα. Γυρίζω σελίδα σε 14 λοιπόν, 59 πίπερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 61 μίλτερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 62 δική μου υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 63. Bradburn Chan υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64. Α, καλύπτεται αυτή. 65 λοιπόν, 65 λοιπόν, Μιλντερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66, οντί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 15. 67. Πίπερ υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτει τότε του κύριου Όντι. 69 πάλι Όντι υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 Όντι υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 Bradburn Czarnek υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ας επαληθεύσουμε παράγος 16 71 Κλείνω την ψηφοφορία. Εγκρίθηκε 15, κατά, 15 ε, υπέρ δηλαδή. 73 Γκάιερ, 72 συγγνώμη Γκάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτει τότε 73, αλλά ψηφίζουμε την 74 δική μου, που είναι ασύμβατη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 75, ότι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 15, 77, οντί, με προφορική τροπολογία του Λαϊκού Κόμματος, υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα επαληθεύσουμε, 77. Πέρας. Απερίφθη 12-15. Ψηφίζουμε τώρα την αρχική τροπολογία. Υπέρ. Έχουμε απορρίψει την προφορική τροπολογία του Λαϊκού Κόμματος. Γι' αυτό τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο της τροπολογίας. Ψήφι υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτό. 78 Μπράντμπουρ εκεί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 Γκάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 Πίπερ υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 81 Γκάιερ υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 82 Σόντεργαρτ Ντε Ναι Γέννη, ορίστε είναι για την 82. Αρχικά είχα ταχθεί υπέρ της τροπολογίας Σόντεργαρτ και Ντε Γιόγκ και γι' αυτό είχα βάλει συν. Νομίζω όμως ότι τακτικά δεν θα μας εξυπηρετήσει και γι' αυτό αλλάζω άποψη. Ωραία. 82 Σόντεργαρτ και με αρνητική τοποθέτηση του συγητού Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, θα χρειαστεί παρήθευση. Είναι πολύ δύσκολο να κρίνει κανείς από την έδρα του προέδρου. 82 λοιπόν. Ε. Λίγη ψηφοφορία. Α, μάλιστα. 20 υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνεται επομένω. Παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια, ψηλά και καθαρά. 83, 83 μάλλον, Γκάιερ. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 84 γκάι. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 αυτή εκπίπτει γιατί έχει ψηφιστεί η σχετική συμβαστική 86 επίση, διότι εγκρίθηκε η 2. 87 δική μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 της κ. Μακοβέη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 89 ντελάνγκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ακολουθεί η σελίδα 16 Η δική μου τροπολογία 90, όπου ζήτησε ψηφοφορία κατά τμήματα το Λαϊκό Κόμμα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε τμήμα 2 της 90. Πέρας. εγκρίνεται 14-13 91 δική μου υπέρ κατά αποχές ας το επαληθεύσουμε 91 ηλεκτρονική επαλήθευση Α, ναι, δεν θα ψηφίσω εγώ. Κλείνω την ψηφοφορία. 17 υπέρ 10 κατά. 92 υπέρ υπέρ. Αυτή εκπίπτει όμως. Η 93 επίσης. Για την 94 έχουμε ψηφίσει τη σχετική συμβαστική τροπολογία. Η 95 καλύπτεται επίσης από την συμβαστική τροπολογία και καταλήγουμε στην 96. Bradburn Τσαρνέκη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη σελίδα 17. Τροπολογίες 97, 98 και 99 ας ψηφιστούν όλες μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι ξεχωριστά λοιπόν 97 ήταν αυτή. 98 Μακοβέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 δική μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 Γκάιερ Μίλτερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 Μπράτβον Τσαρνέκη υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. 101. Κλείνω την ψηφοφορία. 16 υπέρ 11 κατά. Νομίζω μπορούμε από 102 έως 110 συμπεριλαμβανομένων να τα ψηφίσουμε όλα μαζί, όλες μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Όλες λοιπόν αυτές απορρίπτονται. 111 Γκάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 Πίπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, μάλιστα, ε, ηλεκτρονική πολίτηση 112 αρχίζει η ψηφοφορία τέλος απερίφθη με 12 υπέρ 15 κατά μάλιστα πιο μικρή διαφορά από ό,τι μου φάνηκε στην αρχή τώρα 113 δική μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται 115 γκάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 πάλι γκάι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 πίπερ συμβατή με την 116 υπέρ της 117 κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 πίπερ υπέρ 119. Α, έχει αποσυρθεί. και Πίπερ, είστε παρόν. 119 έχει αποσυρθεί. Όχι. Άρα πρέπει να ψηφιστεί. Καλά λοιπόν. 119. Πίπερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη γιατί είχα τη λάθος πληροφορία. 120 γκάιερ υπέρ κατά. Αποχές. Οκ, okay, εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 122 Παναγιώτοβα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 123. Bradwood Τσανίκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124. Αυτή εκπίπτει λόγω της συμβαστικής 2. 125 δική μου υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 126 όντι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 Μακοβέ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 128. Μπράτμπορν Τσαρνέκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129. Κάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130. Παναγιώτοβα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131. Πίπερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132. Παναγιώτοβα υπέρ. Κατά. αποχέεις; Εγκρίνεται και αυτή. Σελίδα 19. Να, πω, να πιω και μια γουλιά νερό. Παράγραφος 66, 133, Μπράτμον Σανέκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134, Πίπερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Τροπολογίες 135, 36, 37, 38. Αυτές καλύπτονται από τη συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, ε, τροπολογία 140, Σόντεργαρτ, υπέρ, Κατά. Επαλήθευση παρακαλώ. 140. Το Λαϊκό Κόμμα φαίνεται να έχει μία ψήφο παραπάνω από όσες δικαιούται. Ωραία, λοιπόν, τότε λίγη η ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Α, ισοψηφία. 14 υπέρ, 14 κατά. Απορρίπτεται. Κρίμα. Κρίμα, Σόντεργαρντ. 141 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 142. Καλύπτεται όμως από την 4 συμβαστική. 143. Μπραντ Μπορντσανέκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 γκάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 δική μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147, 148, 149 μαζί. Καλύπτονται από τη συμβαστική 5. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 150 πράγματα και έτσι ανήκει καταπέπτουν γιατί έχει εγκριθεί συμβαστική. 151 δική μου. Υπέρ και πριν κατά αποχές εγκρίνεται. 152 είναι γλωσσική και δεν την ψηφίζουμε. 153 δική μου και πάλι δε. Κατά. Εποχές ε, εγκρίνεται. 154 επίσης γλωσσική. 155 της κυρίας Μακοβέη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στη 21. Παραγραφός 88, συγγνώμη. 156 υπέρ της Παναγιώτοδο, Παναγιώτοβα. Κατά αποχές εγκρίνεται. 157 Μακοβέ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 158, 59 και 60 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ελέγχουμε τις τροπολογίες αυτές ηλεκτρονικά 158, 59 και 60. Πέρας. 14 υπέρ, 13 κατά εγκρίνεται. 161 υπέρ, με το κύριο Πίπερ, υπέρ κατά, άποχες. Και πάλι εδώ είναι μικρή διαφορά και θέλει έλεγχο. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, ηλεκτρονικά η επαλήθευση την 161. 14 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 162. Με προφορική τροπολογία του κυρίου Μολντερ, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 163. Γκάιε, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 164 γκάιερ υπέρ, κατά, αποχές, γκρίνεται. 165 μακοβέ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 166 γκάιερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 167 γκρέσλι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 168 γκάιερ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 169 Νόλβερ, με την προφορική τροπολογία πέρας Σόντεργατ και Γιόγκ. Υπάρχει μια πρόταση για συμβιβαστική υπαριθμών 6, αλλά πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Σόντεργατ αν συμφωνεί με το συμβιβασμό αυτό. Διαφωνείτε με το συμβιβασμό? Όχι. Εντάξει, εντάξει, ψηφίζουμε. 2,46 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 2,47. Σέντερ Γιόγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 248 των ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 249 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ερχόμαστε στην Επιτροπή Δημοσιοελευθεριών ΛΥΜΠΕ, ένα της ΛΥΜΠΕ υπέρ, κατά, άποχες, έγκρινεται. 2 ΛΥΜΠΕ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 3 και 4 τις λείπει μαζί κατά αποχές εγκρίνεται 2.50 Γκάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.51 Γκάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται